Άρχεται η συνεδρίαση. Όπως ξέρετε, το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα είναι η ψηφοφορία για την αίτηση κατεπήγοντος πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου τροποποίηση του κανονισμού